Okay, dear colleagues, I think we can continue. We are at item 10, implementation of the UN Και συνεχίζουμε με το θέμα της σύμβασης για τα άτομα με αναπηρίες και τα συμπεράσματα της παρατηρήσεις της Αντίστοιχης Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών. Η κυρία Χάουταλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και με την άδειά σας θα σημειώσω ότι η ολίγοι παριστάμενοι δεν υποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τα άτομα αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σχέδιο λοιπόν αυτό γνωμοδότης προσπάθησα να συλλέξω σημαντικά ζητήματα για το πώς η δουλειά μας και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής μας σχετίζονται με τα δικαιώματα των ε, ατόμων με αναπηρία και τη σχετική σύμβαση των ΗΕ. Εθνών. Κάποιοι συνάντητε έχουν καταθέσει τροπολογίες. Ως συγγήτρια τι καλωσορίζω και θέλω να επισημάνω ότι είναι η κυρία Τέβας Φεραγκούτ, Γκόμες Μαστάλκα, Ζαμπάτσκι, Κόσα. Οι τροπολογίες, 31 τον αριθμό, εν γέννη, βοηθούν την γνωμοδότηση, της δίνουν μεγαλύτερο βάθος και ανάλυση. Στην ε, Αθήλυνα αρμόδια επιτροπή, κυρία Στίβενς ως αρμόδια πιστεύω θα συνεργαστεί θα έχει πολύ καλή συνεργασία. Γενικά έχουμε πολύ καλή συνεργασία στην υπόθεση αυτή μεταξύ των επιτροπών. Από τις 31 ε, λοιπόν ε, τροπολογίες όλες προσπαθούν να ενισχύσουν το μήνυμα της ε, πρότασής μας και δεν βλέπω καμία δυσκολία. Ε, θα τις δεχθώ όλες τροπολογίες, συμβαστικές δεν θα έλεγα ότι θα είναι, γιατί τις θεωρώ όλες τις προτάσεις των συναδέλφων ως συμβολή στο κείμενο. Τα δικαιώματα λοιπόν των ατόμων με αναπηρίες και η Σύμβαση των Εθνών. Αυτά από μένα δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι θέλουν να δώσουν κάποιες ε, Εξηγήσει για το πνεύμα των τροπολογιών του εάν κάποιο άλλο θέλει το λόγο. Πριν κάνουμε την διαθέτηση των κειμένων για να έχουμε μια καλή γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Όντως, λέει ο Πρόεδρος, τώρα είναι η ώρα να λάβουν οι συνάδελφοι το λόγο για τα σχόλιά τους. Δεν βλέπω κανείς να σηκώνει το βλέμμα του. Άρα φαίνεται πως δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν. Και ευχαριστώ την κυρία Χάουταλα για την παρουσίασή της. Έχουμε ολοκληρώσει έτσι το σημείο 10. και θα συνεχίσουμε με την ανταλλαγή απόψε με τον Επίτροπο Χίλ για τις αναφορές αναχώρα στις 4.30 άλλα 15 λεπτά διάλειμμα λοιπόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Είμαστε εδώ για να ανταλλάξουμε απόψεις με τον Επίτροπο Χίλ για τι εκθέσεις αναχώρα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο Πρόκειται για μια κοινή συνεδρία των Επιτροπών Γιούρια, Εκον και Τάξε. Είναι παρόντες και οι τρεις πρόεδροι. Γίνεται αυτή η κοινή συνεδρίαση γιατί το ζήτημα αυτό εντάσσεται στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Γιούρη. Εταιρικό δίκαιο δηλαδή. Καλώς ήλθατε κύριε Επίτροπε. Να καλωσορίσω τον ε, κύριο Γκουαλτιέρη, πρόεδρο τη Επιτροπή ΕΚΟΝ. Να καλωσορίσω και τον κύριο Αλαλαμασού, πρόεδρο τη Επιτροπή ε, ΤΑΞΕ. Καλώ ήλθατε. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και επειδή και ο χρόνος του Επιτρόπου είναι περιορισμένος, πρέπει να φύγει στις 6 παρατέταρτο. Να δώσω καταρχάς το λόγο στον κύριο Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που δεχθήκατε να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων με τον Επιτροπό Χίλ σχετικά με τις εκθέσεις αναχώρα στο πλαίσιο μιας κοινή συνεδρίασης των Επιτροπών Εκον Να καλωσορίσω και εγώ τον πρόεδρο τη Επιτροπή Τάξη, τον κ. Λαμασού και φυσικά και τον Επιτρόπο Χιλ. Ήδη έχετε καταθέσει την πολύ αναμενόμενη πρότασή σα για τι εκθέσει αναχώρα στην Ολομέλεια τη προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Θα, ε, έχετε υπόψη σας ότι ήταν πολύ θετικό ο αντίκτυπο η απήχηση αυτή τη πρόταση, που είναι ένα θετικό βήμα προ την ενίσχυση τη εταιρική διαφάνεια στον τομέα τη φορολογία. Πράγματι, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και στο σημερινό πολιτικό πλαίσιο μετά τις αποκαλύψεις ε, των Panama Papers. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ του Κοινοβουλίου ήταν στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις αναχώρα. Είχαμε πρώτα την οδηγία κεφαλαιοακών απαιτήσεων για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τα καταθέσαμε τροπολογίες στην οδηγία για το δείγμα των μετόχων και πιο πρόσφατα στη δική μας έκθεση πρωτοβουλία ζητήσαμε περισσότερη φορολογική διαφάνεια και συντονισμό για, μια, ε, για οριζόντιες εκθέσεις αναχώρα σε όλους τους τομείς. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ σημαντική στιγμή. Επικροτούμε το γεγονός ότι διευρύνθηκε η πρόταση αυτή οι εταιρείε δηλαδή που έχουν θηγατρικέ σε φορολογικού παραδού θα πρέπει να αναφέρουν πλήρω για τι δραστηριότητε που ε, αναπτύσσουν σε αυτέ τι χώρε και τώρα περιμένουμε βέβαια να ξεκινήσουμε και εμείς το νομοθετικό μας έργο για να ενισχύσουμε την περαιτέρω και να βελτιώσουμε την πρόταση αυτή, ιδίως σε ό,τι αφορά ε, τη δημοσιοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και με απότερο στόχο να έχουμε ένα πλήρες σύστημα εκθέσεων αναχώρα για όλες τις φορολογικές δικαιοδοσίες και για την εφαρμογή των κανόνων που είναι εφαρμοστές αυτή τη στιγμή στις τράπεζες σε όλες τις πολυεθνικές και να υπάρχει δυνατότητα επέκταση του πεδίου εφαρμογή αυτή τη πρόταση για να είναι πιο αποτελεσματική και να καλύπτει περισσότερε εταιρείε. Βέβαια, θα δούμε, θα έχουμε ε, και εμεί ε, συμμετοχή σε αυτή την νομοθετική διαδικασία. Σίγουρα όμω θα έλεγα ότι η σημερινή στιγμή είναι ιστορική, το ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε εδώ. Ε, οι τρεις επιτροπές από το έργο μας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι τώρα. Ε, να δώσω το λόγο στον Αλέν Λαμασού να μας κάνει και αυτός μια εισαγωγή. Ευχαριστώ Πρόεδρε που δεχτήκατε να γίνει αυτή η ακρόαση. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο Χίλ που ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ο Επίτροπο δεν έρχεται παρά μόνο αν βρίσκεται ενώπιον τριών επιτροπών. Μόνο μπροστά σε τρει επιτροπέ θέλει να μιλήσει. Μεταξύ τα των πολλών νέων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα περισσότερα βεβαίω είναι κακά νέα. Και αυτό που θα μα απασχολήσει ε, όμως είναι ένα καλό μελλοντικό νέο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω από κάποια κράτη-μέλη ε, έχουν ξεκινήσει έναν αγώνα που θα κερδίσουν κατά τη φοροδιαφυγή των πολυεθνικών. Μετά το LuxLeaks, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιούργησε μια ειδική προσωρινή επιτροπή που υιοθέτησε διάφορες συστάσεις μέσω στην Ολομέλεια, μέσω της Ολομέλειας, ε, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή ΕΚΟΝ, που επίσης υιοθέτησε κάποιες συστάσεις και που αφορούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γενικό επίπεδο το, οι ειδικέ αναχώρα εκθέσεις αφορούσαν αυτές τις συστάσεις. Θέλουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Δεν θέλουμε να αφορά η διαφάνεια μόνο τις φορολογικές αρχές και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ακολουθεί σε αυτή τη διάθεση για διαφάνεια. Όπως είπε ο κ. Γκουαλτιέρη, βασιζόμαστε στα προηγούμενα που έχουμε ε, με τη συνεμπειρία που έχουμε συσσωρεύσει με τις τράπεζες και με τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ε, κάναμε ακροάσεις στην τάξη και ομολόγησαν ότι επειδή δημοσιοποίησαν διάφορα οικονομικά στοιχεία, αυτό δεν σημαίνει ότι επλήγει ο ανταγωνισμός του σε σχέση με, Αμερικαν... με ανταγωνιστές από την Αμερική ή την Κίνα. Εμείς ήρθαμε σε επαφή με διάφορες πολυεθνικές, αμερικανικές κυρίως, που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία και θέσαμε το ερώτημα, είσαστε έτοιμες για αυτή την, ε, τις, τις εκθέσεις ε, αναχώρα, τις ειδικές ε, εκθέσεις αναχώρα και είσαστε έτοιμοι να δημοσιοποιήσετε διάφορα λογιστικά στοιχεία που σας ζητάνε οι εφορίες. Πάνω από τις μεσές είπαν ναι. Παραδείγματο χάρη, οι εταιρείε που κατασκευάζουν κινητά τηλέφωνα. Υπάρχουν δύο μεγάλες εταιρείε. Αρκεί ο ένας από τους δύο αυτού εταίρου να πάρει την πρωτοβουλία να δημοσιοποιήσει αυτά τα στοιχεία, ούτως ώστε να ακολουθήσει υποχρεωτικά και ο άλλος να κάνει το ίδιο. Γιατί αλλιώς θα χάσει τη φήμη του ότι είναι σοβαρή εταιρεία και θα θεωρηθεί κακός φορολογούμενος. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή η συζήτηση και αυτή η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυρίως ε, σημαντικά τα συμπεράσματα ε, της ε, έκθεσης αυτής που έκανε η Επιτροπή και της μελέτης αντικτύπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και αυτά. Σας ευχαριστώ και τώρα θα ήθελα ο Λόρδος Χιλ να κάνει την παρουσίασή του. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Σας ευχαριστώ που μαζευτήκατε εδώ και οι τρεις επιτροπές. Χαίρομαι που είμαι εδώ ενώπιόν σας και που έχω την ευκαιρία να σας πω επίσημα ότι εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά που κάνατε στον τομέα αυτό. Εγώ έπαιξα ένα μικρό ρόλο, συμμετείχα λίγο, άλλοι κάναν πολύ περισσότερα, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που είχα την ευκαιρία να σας παρουσιάσω αυτή την πρόταση. Όπως είπε ο κύριος Γκουαλτιέρη, οι αποκαλύψεις από τα Panama Papers φυσικά έχουν δώσει νέα ορμή στη συζήτηση για τις τη φορολογία. Και η πρόταση για τις ειδικές της τάσης έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από το Panama Papers και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα φορολογικής μεταρρύθμισης όπου νομίζω ότι όλοι μας έχουμε σημειώσει πολύ πρόοδο. Ε, με τη συνάδελφο Μάρκετ Φεστέρ νομίζω ότι ασχοληθήκαμε με τις με την επιλεκτική φορολόγηση. Ο Πιέρ Μοσκοβισή έχει προωθήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ε, σε χρόνο ρεκόρ ε, για την αυτόματη ανταλλαγή των φορολογικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών. Έχουμε ε, υπογράψει συμφωνίες για τη φορολογική διαφάνεια, για τα μερίδια με το, με το Λιχτενστάιν, την Ανδρό, Σαμαρίνο, την Ελβετία και θα κάνουμε πολύ περισσότερα. Και διεθνώς συνεργαζόμαστε στενά με τον ΩΣΑ και τον G20 για να προωθήσουμε την ε, παγκόσμια καλή διακυβέρνηση στο χώρο το φορολογικό. Η πρόταση περασμένη εβδομάδα για τις ειδικέ αναχώρασει τάσει συνάδουν όλη αυτή την προσπάθεια και όλη αυτή την προσέγγιση για μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά όχι μόνο. Και κάτι παραπάνω εξασφαλίζουν. Απαιτεί από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές του κόσμου να δημοσιεύουν βασικές πληροφορίες για τους φόρους που πληρώνουν και πού πληρώνουν αυτούς τους φόρους. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξή. Θα είμαστε η πρώτη δικαιοδοσία στον κόσμο που θα πετύχει κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι ορισμοί είπαν ότι οι φορολογικές πληροφορίες δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται, ότι θα πρέπει να αφορά μόνο ε, τις φορολογικές αρχές. Έχω να σας απαντήσω ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια μπορεί να εξασφαλίσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, να μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε το αν έχουμε τη σωστή νομοθεσία και το αν υπάρχουν παραθυράκια τα οποία θα πρέπει να κλείσουν. Νομίζω ότι θα ενθαρρύνει τις εταιρείε να σκεφτούν αν δρούν ε, σωστά μακροπρόθεσμα υπέρ των μετόχων τους, ε, αν είναι και αν έχουν μια σωστή στάση, νομίζω είναι καλό για τις ε, δουλειές τους, για τις επιχειρήσεις. Καλό είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη στον επιχειρηματικό κόσμο. Ελπίζω ε, επίσης ότι θα μας βοηθήσει να εστιάσουμε σε βασικά θέματα που είναι πώς κρατάμε την ισοτιμία, πώς προστατεύουμε την ανταγωνιστική θέση της, ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης. Να θυμηθούμε κάτι όλοι μας. Εκτιμάται ότι οι πολυεθνικές μπορούν να πληρώσουν 30% ε, λιγότερο από τις μικρότερες ε, εταιρείες που λειτουργούν μόνο σε μία χώρα. Είναι σωστό αυτό. Είναι δυνατό να είναι σωστό από τη σκοπιά του ανταγωνισμού. Και πώς είναι δυνατόν ε, να είναι δίκαιο και ισότιμο. Δεν πρέπει να συμβαίνει έτσι. Οι μικρότερες εταιρείε, οι οποίες δεν μπορούν να μετακινήσουν τα κέρδη τους ή μπορούν να έχουν έξυπνες φορολογικές συμβουλές να έχουν αυτό το φορολογικό το ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τι πολυεθνικέ. Αν κάποιε εταιρείε πληρώνουν λιγότερου φόρου, αυτό σημαίνει ότι κάποιε άλλε πληρώνουν περισσότερου. Σημαίνει ότι οι μικρότερε εταιρείε πληρώνουν για λογαριασμό των πολυεθνικών. Αυτά που δεν πληρώνουν οι πολυεθνικέ. Εγώ είμαι υπέρ των επιχειρήσεων, υπέρ του ανταγωνισμού, αλλά ο ανταγωνισμό που θα ήθελα να υπάρχει είναι ανταγωνισμό για τι υπηρεσίε, για τι τιμέ, για την ποιότητα, για την καινοτομία των προϊόντων και όχι για να υπάρχει έτσι, μια δημιουργικότητα στις φορολογικές συμβουλές. Εάν θέλουμε λοιπόν μεγαλύτερη και πετύχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, ε, θα εξασφαλίσουμε τις εξής αρχές. Καταρχάς, συνέπεια με τη διεθνή προσπάθεια που γίνεται από τον ΩΣΑ ε, και που έχει επικυρώσει τον G20, θα βασιστούμε στις βασικές μεταρρυθμίσεις που είναι εξελίξη ε, και που ξεκίνησε ο Πιέρα Μοσκοβισή, θέλουμε να καλύψουμε όλες τις ε, πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, όχι μόνο τις ευρωπαϊκές, και θέλουμε βεβαίως να είμαστε αναλογικοί σε αυτό που κάνουμε, ούτως ώστε να μην υποσκάπτουμε τη θέση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ε, απέναντι στους παγκόσμιους ανταγωνιστές τους, ούτε να επιβαρύνουμε τις μικρομεσαίες ευρωπαϊκές, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που κλασικά δραστηριοποιούνται μόνο σε μια χώρα. Αυτό που θέλει λοιπόν η πρότασή μας να πετύχει είναι ότι στο μέλλον οι μεγάλες πολυεθνικές με ετήσια έσοδο ε, πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ ετησίω θα πρέπει να ε, δημοσιοποιούν πληροφορίε σε διάφορου βασικού τομεί. Θα αφορά ε, γύρω στι 6.000 πολυεθνικέ, ευρωπαϊκέ και μη ευρωπαϊκέ και υπ' αυτή την έννοια ε, ξεπερνάει τις προηγούμενες προτάσεις που αφορούσαν μόνο τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό είναι σημαντικό, νομίζω, για λόγους ισοτιμίας, αλλά επίσης γιατί θέλω να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που δημιούργησαν ανησυχίε για τις μη ευρωπαϊκές πολυεθνικές που πληρώνουν ε, ελάχιστους ή καθόλου φόρου σε, χώρε στις χώρες όπου παράγονται τα κέρδη. Στο μέλλον λοιπόν με αυτές τις ε, ειδικέ αναχώρασεις τάσεις θα δημοσιεύονται η φύση των ε, δραστηριοτήτων τους, ε, το προσωπικό, ο τζίρος, το κέρδος πριν τη φορολογία, ο φόρος που πληρώνουν την κάθε χρονιά και το συσσωρευμένο, τα συσσωρευμένα έσοδα. Επίσης, οι πολυεθνικές θα πρέπει να αναφέρουν ε, το συνολικό φόρο που πληρώνουν εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, θα πρέπει, αποφασίσαμε μάλλον, ότι αν οι φόροι πληρώνονται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρε όπου δεν γίνονται σεβαστά τα διεθνή πρότυπα για του φόρου, τότε οι πολυεθνικέ θα, πρέπει, θα πρέπει να δημοσιεύουν λεπτομερή στοιχεία με τον ίδιο τρόπο που τα δημοσιεύουν σε περίπτωση που πληρώνουν στην Ευρώπη του φόρου. Όλε αυτέ οι πληροφορίε θα μα δώσουν σαφή εικόνα για το αν μια μεγάλη πολυεθνική πληρώνει φόρου και αν πληρώνει εκεί που παράγεται το κέρδο, Οι πληροφορίε θα πρέπει να δίδονται για πέντε χρόνια στην ιστοσελίδα τη εταιρεία και οποιοδήποτε ενδιαφέρεται θα μπορεί να δει τα στοιχεία αυτά, πού πληρώνουν του φόρου δηλαδή πολυεθνικές και αν υπάρχει ισοτιμία και ισότιμη μεταχείριση όλων των εταιριών. Για να μην είναι σε μειωθική θέση οι ευρωπαϊκέ εταιρείε, οι κανόνε αυτοί θα αφορούν και τι θηγατρικέ των μη ευρωπαϊκών πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, καθώ και τι μεγάλε ευρωπαϊκέ πολυεθνικέ. Ε, οι ευρωπαϊκές τράπεζες ε, συμμορφώνονται ήδη με το ειδικό καθεστώς ε, διαφάνειας για τις τη κεφαλαϊκή επάρκεια κτλ. Δεν θα αλλάξει τίποτα εδώ. Οι μεγάλες τράπεζες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δρασιοποιούνται στην Ευρώπη όμως θα πρέπει στο μέλλον να δημοσιεύουν ειδικέ αναχώρα εκθέσεις. Ετοιμάζοντα την πρόταση, κοιτάξαμε του κανόνε που ισχύουν για τι τράπεζε, για την εξορρυπτική βιομηχανία και τι ιδέε που συζητιώνται στο Κοινοβούλιο για τα, την οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων και θέλουμε μια ε, ισορροπημένη προσέγγιση που να μην είναι κατά τη ανταγωνιστικότητα, αλλά ε, φιλόδοξη ό,τι αφορά τη φορολογική διαφάνεια. Μια ερώτηση που μα θέσαμε. Γιατί ε, δεν θέλουμε λεπτομερή νούμερα εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, γιατί η μελέτη αντικτύπου μας έδειξε ότι αν οι εταιρείε εκτός Ευρώπης δεν δημοσιεύουν τις χίλιες πληροφορίες, ε, τότε θα θέτουμε σε μειονεκτική θέση τι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Καταρχά, οι εμπορικοί ανταγωνιστέ του θα έχουν πληροφορίε για αυτέ που δεν θα έχουν ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, όμω για του ανταγωνιστέ και οι εταιρείε μπορεί να είναι σε ευάλωτη θέση, μπορεί να ε, φορολογηθούν δύο φορές εντός και εκτός Ευρώπης. Εφαρμόζοντας αυτή την ε, ε, νομοθεσία με, ε, σε εταιρείε πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ τζίρο, θα καλύψουμε περίπου όλες τις πολυεθνικές, το 90% περίπου. Αυτό συμφώνησαν και στο G20, στο BEPS, στο NOSA. Καλύπτουμε τις εταιρείε που έχουν την ικανότητα να κάνουν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό όλες οι εταιρείες οι οποίες ε, διερευνώνται ε, για κρατικές ενισχύσεις ε, κτλ. χωρίς να βαραίνουμε τις μικρότερες επιχειρήσεις που αποκλείεται να εμπλέκονται σε τέτοιε προσπάθειε φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή. Άκουσα τι απόψει διαφόρων ενδιαφερομένων και το αποτέλεσμα νομίζω είναι μια πρόταση απλή αναλογική και θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε την λογοδοσία, θα μας βοηθήσει να έχουμε μια πιο σοβαρή συζήτηση για το που πληρώνουν φόρους οι εταιρείε και το δίκαιο που διέπει την, νομοθεσία, την φορολογία, δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Τώρα θέλω να συνεργαστώ στενά με το Κοινοβούλιο και με τα κράτη-μέλη, ώστε να συμφωνηθεί η πρόταση αυτή, να περάσει αυτή η πρόταση και να εφαρμοστεί βεβαίως. Thank you very much, Commissioner. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ξεκινήσουμε τον γύρο των ερωταπαντήσεων τώρα. Η Επιτροπή Γιούρη έχει την προτεραιότητα, αν κατάλαβα καλά, μπορεί να ξεκινήσει δηλαδή ένας βουλευτής επιτροπής αυτής. Θα έχουμε τέσσερις ερωτήσεις, διάρκεια σε κάστη δύο λεπτών. Και θα υπάρξει και μια δεύτερη δέσμη ερωτήσεων θα παρακαλέσω τους συναδέλφους ε, να μην εξαντλούν το χρόνο τους για να μην χρόνος και για τους υπολείπους. Θα ζήσει, θα επιζήσει ο Επίτροπος ε, ε, και μην ακούσει από όλους να τον ευχαριστούν για την καλή δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Λοιπόν, κυρία Ρέγνερ είναι η πρώτη. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας, κύριε Επίτροπε. Ξέρω ότι χάρη στις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις πολυάριθμες εκθέσεις, Dot, Tally και άλλες ε, με πρώτα βέβαια την έκθεση για τα δικαιώματα των μετόχων έχουμε φτάσει στην πρόταση που κατατέθηκε ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα βεβαίως θα αναφερθώ στο όριο γιατί κάνατε αναφορά σε 750 εκατομμύρια κύκλο εργασιών δεν είναι πολύ φιλόδοξο αυτό ξέρουμε ήδη τι κάνει ο ΩΣΑ πολύ ωραία, ωραίες προσπάθειες αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προχωρήσει έτσι περαιτέρω το αναφέρατε και νωρίτερα ότι η οδηγία για, το, για τα λογιστικά, για τη διαφάνεια ήδη δίνουν παραδείγματα και βεβαίως κάποιοι μπορούν να λένε αν δεν χρειάζεται να πάμε τόσο ε, μακριά. Γιατί δεν παίρνετε λοιπόν αυτό ως παράδειγμα στο εταιρικό δίκαιο. Έχουμε μικροεπιχειρήσεις, ε, μεσές, ε, μικρές και μεσές επιχειρήσεις και μεγάλες. Τώρα θέλετε να εισαγάγετε και μια νέα κατηγορία των υπερμεγεθών εταιριών. Έχει νόημα αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ απλό. Μπορείτε απλώ να βάλετε σαν κανόνα ότι οι επιχειρήσει πληρώνουν φόρο εκεί που ε, αποκομίσουν το κέρδο. Κυρία Νίμπλερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Μια πρώτη αξιολόγηση και μου επιτρέψετε και μια ερώτηση ω προ την αξιολόγηση. Η πρόταση πιστεύω εξισορροπεί ικανοποιητικά την ανάγκη για διαφάνεια και περισσότερη φορολογική δικαιοσύνη αφενός και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που επίση θα πρέπει να διαφυλαχθεί αφετέρου. Τα καταφέρνει λοιπόν αυτά, άρα την αξιολογούμε θετικά. Έχω μία ερώτηση και σας παρακαλώ να δώσετε περισσότερες εξηγήσει στη δήλωσή σας αυτή. Στο πλαίσιο του ΣΑΙΠΑΤΕ είπατε, ε, υπάρχουν πιο φιλόδοξοι, πιο φιλόδοξες προσεγγίσεις, λιγότερο φιλόδοξες προσεγγίσεις. Εξηγήστε το μας αυτό και πείτε μας επίσης η δική μας νομοθεσία μέσα στον όλο διάλογο του σε επίπεδο τι θέση λαμβάνει. Ευχαριστώ Κοφεράτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, Επίτροπε. Δύο ερωτήσεις να σα κάνω, πολύ γρήγορες. Πρώτον, για ποιο λόγο το οικοδόμημα αυτό τελικά είναι πολύ πιο μικρό από το οικοδόμημα που φτιάξετε για τις τράπεζες. Εάν δούμε το κατόφλι που βάλατε, τις πληροφορίες που μπαίνουν και το πεδίο εφαρμογή. Έχουμε μία λύση για τις ε, επιχειρήσεις, σαφώς λιγότερο φιλόδοξη από αυτή που έχουμε για τις τράπεζες. Πάντα εσείς μας λέγατε ότι μετά από την ε, μελέτη σκοπιμότητας που κάνατε, μήνες σας πήραν το κάνετε αυτό το κείμενο, ε, θα φτάνετε σε ανάλογες λύσεις, τράπεζες και επιχειρήσεις. Όμως με θλίψη παρατηρώ ότι κλείνοντας ε, αυτή τη ε, μελέτη σκοπιμότητας φτάσατε σε μία λύση χωρίς να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό για τις τράπεζες και δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν προκύπτει το γιατί. Δεύτερον, είπατε ότι αυτή η νομοθεσία θα είναι πάρα πολύ σημαντική για τους μετόχους. Και εμείς είμαστε πεπισμένοι γι' αυτό. Γιατί... Γιατί προτείναμε με μία ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο ένα σενάριο πολύ πιο φιλόδοξο από το συμπέρασμα στο οποίο φτάσατε εσείς στην οδηγία για τους μετόχους. Δηλαδή, αν υπάρχει ήδη ένα κείμενο, το οποίο έχει ψηφιστεί ήδη, αν υπάρχει ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τους ε, μετόχους για να γνωρίζουν ποια είναι η φορολογική πραγματικότητα της ε, επιχείρησης αυτής γιατί να μην χρησιμοποιήσετε αυτή την οδηγία λοιπόν που έχουμε ψηφίσει, αντί να φτιάξετε κάτι τελείω καινούριο, το οποίο θα έχει δύο μειονεκτήματα. Πρώτον, μπορεί να ακροτηριάσει την οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων πρώτον και δεύτερον, ούτως ή άλλως για να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα θα χρειαστεί χρόνο, θα πάρει χρόνο όλη αυτή η ιστορία. Πολύ πιο απλό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε την οδηγία που ψήφισε το Κοινοβούλιο για τα δικαιώματα των μετόχων. Γιατί δεν το κάνατε. Uh, η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που ήρθατε στην Επιτροπή μας και θέλω να σας ευχαριστώ για τον τρόπο της δημόσιας ενημέρωσης που επιλέξατε. Εξήγησατε και τους λόγους. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω καταρχάς για τα ε, όρια στην ε, πατρίδα μου τη Φιλανδία αισθανθήκαμε με το δημόσιο διάλογο που έγινε βέβαια και την ε, ντροπή της συζήτησης αν επρόκειτο για 100 ή 200 εκατομμύρια για τις μεγάλες ε, επιχειρήσεις οι οποίες μάλιστα είχαν καταγραφεί και ως πρώτης ποιότητας. Θα ήθελα λοιπόν αυτό το όριο που θα οριστεί να εξυπηρετεί πραγματικά το δημόσιο συμφέρον. Και η πρώτη πρόταση που είδαμε σε σχέση με την φορολογική πληροφορία σε ενοποιημένη μορφή προς τον υπόλοιπο κόσμο που φάνηκε θα έλεγα κάπως επίοικος παράλογη γιατί αποκαλύφθηκε βέβαια η με τα έγγραφα του Παναμά. Τώρα βλέπουμε στο 48GZ ε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κατεψιδότηση πράξης ε, μπορεί να ορίσει κατάλογο για τις περιπτώσεις που παρουσιάζουν τέτοιες δυσκολίε ως προς τη φορολογική κατανομή. Ωστόσο τα κριτήρια είναι πάρα πολύ ασαφή και δεν προκύπτει καν ότι ορίζεται κάποια προθεσμία για να το πράξει. αυτό. Θέλετε να το σχολιάσετε. Ωραία. Ακούσαμε τις τέσσερις πρώτες ερωτήσεις. Ε, Επιτροπή Γιούρη, να απαντήσει ο Επίτροπος. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και για το καλωσόρισμα. Φυσικά επανέρχεται το ζήτημα των ε, κατώτατων ορίων, των κατοφλίων. Και θα σας ε, εξηγήσω τα σχετικά όπως και γιατί Υπάρχει αυτή η διαφορά σε σχέση με τις τράπεζες και στο τέλος τα κριτήρια για τη μαύρη λίστα, τα τεξουσιάδες πράξεις κτλ. Σε ό,τι αφορά τα κατόφλια και αυτό σχετίζεται με το ερώτημα με τον ΩΣΑ και σε διεθνές επίπεδο πώς συνεργαζόμαστε. Η όλη προσέγγιση για μένα εμπνεύστηκε αν θέλετε από την επιθυμία τις μη ευρωπαϊκές πολυεθνικές να ε, μην τις αφήσουμε εκτός ε, και να μην περιουστούμε μόνο στι ευρωπαϊκέ. Υπάρχει νομίζω γενική αίσθηση και διαβάζουμε πολλέ ιστορίε για μη Ευρωπαϊκέ πολυεθνικές που φαίνεται να μην πληρώνουν καθόλου φόρου ή να πληρώνουν ελάχιστου φόρου στην Ευρώπη. Αν στόχος λοιπόν είναι να έχουμε κάτι που θα ισχύει και για τις ευρωπαϊκές και για τις μη ευρωπαϊκές πολυεθνικές και θεωρώ ότι είναι λογικό κάτι τέτοιο, τότε Υπάρχει για εμά ο εξή περιορισμό, αν θέλουμε ισότιμο ανταγωνισμό, ισότιμο πεδίο. Είναι κατά πόσον μπορούμε ή δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε κανόνες και να επιβάλλουμε κυρώσεις έξω εδαφικά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε αμερικανικές εταιρείες που αναπτύσσουν δραστηριότητα στη Σιγκαπούρη, στην Κίνα ή οπουδήποτε αλλού να συμμορφούνται προς τις ίδιες απαιτήσεις που ε, θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό ε, μας καθοδήγησε, αυτό ήταν ο γνώμονας ε, του να έχουμε αυτά τα αναλυτικά, τα μία ομαδοποιημένα στοιχεία και να θετήσουμε αυτή την προσέγγιση. Ό,τι αφορά το κατόφλι, κατανοώ φυσικά τις απόψεις των βουλευτών και τα επιχειρήματά τους και φαντάζομαι ότι όσο προχωράει η νομοθετική διαδικασία θα ε, συνεχίζουμε να ακούμε για το κατόφλιο και κατά πόσο θα ήταν Καλύτερα ένα κατώτερο, πιο μικρό. Εγώ αυτό που θέλω είναι να έχουμε κάτι που θα μας βοηθήσει να ε, καλύψουμε το 90% ε, του των εταιρικών εσών, τις μεγαλύτερες, περισσότερες μεγάλες πολυεθνικές. Ε, αυτό συμφωνεί και με τον ορισμό του ΩΣΑ και νομίζω ότι είναι σημαντικό πάντα για τον ΩΣΑ μιλώντας να Είμαστε φιλόδοξοι και θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι. Με αυτή την πρόταση υπήρξαμε φιλόδοξοι και προχωρήσαμε και πιο μακριά από οποιονδήποτε άλλον ε, μέχρι στιγμής στον κόσμο. Ωστόσο, για να επιτευχθεί μια διεθνή συμφωνία, και αυτό είναι ο στόχο που επιδιώκουμε, είναι λογικό νομίζω στο μέτρο του δυνατού να συμβατίζουμε με κάποιες άλλες πρωτοβουλίε, να δώσουμε εμεί το να λαμβάνουμε τι πρωτοβουλίε και αυτό κάνουμε νομίζω, αλλά να είμαστε συνεπεί. Και νομίζω 750 είναι συνεπέ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι τράπεζε. Μέρος της απάντησης ε, και πάλι είναι ότι θα μπορούσαμε αυτό να το επιβάλλουμε σε ευρωπαϊκές τράπεζες, ε, αλλά όχι ε, άλλες αλλά στόχο στόχος μας είναι, παραλαμβάνω, να ισχύει και για τις μη ευρωπαϊκές. Επίσης, απαιτήσει σε ό,τι αφορά ε, τις ε, τραπεζικές εκθέσεις. Στόχος μας ήταν να αντιμετωπίσουμε προβλήματα χρηματοοικονομικής αστάθειας. Θέλαμε δηλαδή να δοθεί στον κόσμο ε, η απαιτόμενη ενημέρωση για να υπάρχει φορολογική διαφάνεια και πράγματι υπάρχουν ε, κάποιες περαιτέρω πληροφορίες που δίνονται πλέον σε σχέση με το τραπεζικό μοντέλο. Σε ό,τι αφορά την κατεξουσιοδότηση πράξη και τα κριτήρια, δεν υπάρχει προθεσμία. Ο Πιέρ Μασκοβισή νομίζω είπε ότι στόχος του θα είναι να συντάξει μέσα σε έξι μήνες αυτό τη λίστα, αυτόν τον κατάλογο και θεωρεί έτσι νομίζω τουλάχιστον ότι είναι δυναμική η όλη διαδικασία. Υπάρχουν δηλαδή αυτά τα τέσσερα ε, ευραία κριτήρια, θα τα χαρακτήριζα. Και υπήρχαν δικαιοδοσίε, αν μάλλον υπάρχουν δικαιοδοσίε που δεν τηρούν ένα ή δύο από αυτά, ξεκινάμε τη διαδικασία. Χωρί όμω ε, να χρειάζεται, αν μπορεί να αποφευθεί αυτό, να μπαίνουν κάποιοι στη μαύρη λίστα. Αυτή θα είναι πάντως η βάση για τη μαύρη λίστα. Γνωρίζω ε, από τις συνομιλίες που είχαμε τον Πιέρ πόσο θέλει να προχωρήσει αυτό το θέμα. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος θα μπορέσει να σας το εξηγήσει όταν έχει την ευκαιρία. Ευχαριστώ. Χίλ, κύριε Χίλ, ευχαριστούμε και πάμε τώρα στις ερωτήσεις από τους βουλευτές της Επιτροπής των Οικονομικών. Ωστόσο, δεν μπορώ παρά να επισημάνω ότι μια και η δουλειά μας, κομμάτι της δουλειάς μας θέλω ε, στο είναι να συνομιλούμε με τράπεζες, Έχουμε ακούσει πολλές βέβαια διαμαρτυρίες εν γέννη, αλλά δεν άκουσα ποτέ να μας λένε ότι θα τις ε, φέρνει σε ε, δυσμενή ανταγωνιστική σχέση αυτή η πρόταση για τις εκθέσεις ανακράτως. Άρα δεν επιβεβαιώνονται από το κλάδο τον ίδιο αυτή η κίνδυνη που αναφέρεται. Ο κύριος Ροζάτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Και καλώ ήρθατε, Επίτροπε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι θέλουμε να αγωνιστούμε κατά τη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και γι' αυτό αυτή η εφόρμηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του τελευταίου μήνε είναι ιδιαίτερα σημαντική για μα. Βλέπουμε πολλά σημαντικά νομοθετήματα. Φτάνουν μέχρι εδώ στο Κοινοβούλιο. Σήμερα συζητούμε ακόμη ένα σχέδιο προτάσεως για την αποκάλυψη πληροφοριών φόρου εισοδήματος ορισμένων επιχειρήσεων και θηγατρικών. Θα ήθελα λοιπόν να κολοσορίσω αυτή την πρόταση για ένα πιο αποτελεσματικό, διαφανές και ισοδίκιο φορολογικό σύστημα. Για τα μέτρα λοιπόν που θα εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Υπάρχει κάποια πρόθεση να ζητήσετε από τα κράτη-μέλη μία σειρά από συστάσεων ή υποβάλλετε στα κράτη-μέλη μία σειρά από συστάσεων για το πώ θα υλοποιήσουν αυτή την οδηγία. Σε ποιο βαθμό δηλαδή μπορείτε να έχετε υπόψη ενδεχομένω ένα ομοιόμορφο, ένα σύνολο κανόνων, ε, συστάσεων, ακόμη και εξαιρέσεων που θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ακολουθούν σε μια προσέγγιση κατά το μάλλον ή τον ομοιόμορφη ώστε να υπάρξει η νέα, η ίδια προσέγγιση φορολογικά ε, έναντι των επιχειρήσεων και επίσης για τα όρια αυτά που προτείνεται. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι δεν πρέπει να ορίζουμε υπερβολικά υψηλά τον πύχη και πρέπει λίγο πολύ να ακολουθούμε τις προδιαγραφές του ΩΣΑ για τα όρια γιατί δεν μπορούμε να φέρουμε τις επιχειρήσεις μας σε ε, δυσμενή ανταγωνιστική θέση. Αλλά δεν έχουν ε, το, ε, σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι και χωρίς όρια μία επιχείρηση θα μετακινηθεί σε κάποια άλλη δικαιοδοσία προκειμένου να εκμεταλλευτεί ένα άλλο υψηλότερο όριο αφού αυτή η δικαιοδοσία δεν θα καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής οδηγίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό ε, το πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων είναι ισότιμο. Είναι θεμελιώδες αυτό στην Ευρώπη. Είπατε και εσεί ότι όταν είναι υψηλότερο το φορολογικό βάρος για τις επιχειρήσεις κατά 30% καταστρέφονται θέσεις εργασία στην Ευρώπη αφού οι μικρομεσαίες είναι ραχοκοκαλιά τη οικονομία στην Ευρώπη. Ε, είπατε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει για όλες τις χώρες του κόσμου η ε, αναφορά αναχώρα. Μα το εξήγησατε αυτό. Ταυτόχρονα εξηγείτε ότι ενδέχεται να ζητηθεί αναφορά αναχώρα με δημοσίευση σε ε, ειδικέ δικαιοδοσίε, φορολογικού παραδείσου κτλ. Αν λοιπόν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι τέτοιο για ορισμένε χώρε, γιατί όχι και για τι υπόλοιπε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την ερώτηση έχω. Δεν μου φαίνεται πολύ λογικό αυτό που είπατε. Και επίση σε πρακτικού όρου. ο κατάλογος των μη συνεργαζομένων δικαιοδοσιών. Πώς μπορείτε να είστε σίγουρος ότι θα έχει ετοιμαστεί εγκαίρος πριν διατυπωθούν οι απαιτήσει για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και μήπως θα έπρεπε να μπαίνουν σε ένα κατάλογο αυτές οι εταιρείε, ακόμα και οι χώρες, μέχρι όταν αποδεικνύεται ότι έχουν τηρήσει τις προδιαγραφές. Δεν θα ήταν πιο αποτελεσματικό αυτό. Γιατί την αντίστροφη σειρά που επιλέγει η Επιτροπή δεν την πολύ καταλαβαίνω. Ευχαριστώ, Μέστερ Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, που ήρθατε. Είδα την παρουσίαση των νέων κανόνων ε, για, τους, ε, για τη φορολογική διαφάνεια για τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ε, συνδέσατε λοιπόν συγκεκριμένα τα έγγραφα του Παναμά με την αποφασιστικότητα να καταβάλλονται οι φόροι εκεί όπου παράγεται το κέρδος και έτσι η πρόταση θεωρώ ότι πάει λίγο πιο πέρα ακόμα, ζητεί από τις μεγάλες πολυεθνικές να δημοσιοποιούν κέρια σημασία πληροφορίε. Πάντω, εγώ έχω ενημέρωση ότι τα έγγραφα του Παναμά δεν έχουν να κάνουν με πολυεθνικέ τόσο και τι επιθετικέ, λιγότερο υπεστερονόμιμε φορολογικέ του ε, ε κινήσει, αλλά έχουν να κάνουν τα έγγραφα του Παναμά με διαφθορά πολιτικών, ε, ηγετών ακόμη κρατών και κυβερνήσεων προσπαθούν να αποκρύψουν τα περιουσιακά στοιχεία. Ερωτώ λοιπόν, εσείς πώς ακριβώς σκοπεύετε να προωθήσετε τους κανόνες για την εφαρμογή, ε, που θα εφαρμόζονται στις πολυεθνικές για την αντιμετώπιση πιθανών ποινικών αδικημάτων που έχουν αποκαλύψει τα έγγραφα του Παναμά, γιατί δεν βλέπω ακριβώς το συσχετισμό με τη φορολογία των πολυεθνικών. Δεμάση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ, ε, Επίτροπε Χίλ, που είστε εδώ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω και εγώ την ερώτηση του συναδέλφου Κόφαρτ. Δεν βλέπω ακριβώς με ε, ποια είναι η επιλογή αυτή του συστήματος που σας οδηγεί στην απέτηση για τη δημοσίευση ε, για τις εκθέσεις εκεί, εις, βάρος εκείνων που βρίσκονται σε, μαύρο, σε μια μαύρη λίστα ενώ όλοι οι άλλοι δεν έχουν υποχρέωση. Έχετε κάποια νομική πραγματογνωμοσύνη που σας επιβεβαιώνει ότι είναι κάτι τέτοιο αδύνατο ότι το αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει δηλαδή. Και πάντως θα σας έλεγα καλά γλέντια με, την, ε, με, το μαύρο, με τη μαύρη αυτή λίστα γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν με μαύρες λίστες, το 2009 συγκεκριμένα που ξεκίνησαν μεν, μέσα σε δύο-τρεις μέρες είχαν μείνει κενές περιεχομένου, γιατί ε, αμέσω αμέσω υπόθηκε Α, τον Τελαγουέρ των ΗΠΑ γιατί δεν μπαίνει. Η Πορτογαλία επίσης με 78 κράτη στο, στη μαύρη λίστα, ενώ η Γερμανία είχε 0 κράτη στη μαύρη λίστα. Λοιπόν, σας εύχομαι καλά γλέντια στην ε, κατάρτιση αυτού του καταλόγου. Και επίσης υπάρχει μια συγκεκριμένη περίπτωση πολυεθνικών ε, ομήλων και εμεί πρέπει αυτό να το επιβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να ε, δημοσιεύουν τα στοιχεία των, ε, της παραγωγής τους και των κερδών τους. Εμένα ο θείος μου είναι Ιταλός, είναι υποδηματοποιός, κρατάει τα στοιχεία του όλα μέσα σε ένα ντουλάπι, οποτεδήποτε το αισθήσουν πρέπει να τα δηλώσει, πρέπει να τα παρουσιάσει και βέβαια κλαίω όταν βλέπω αυτά τα πράγματα που γίνονται και θεωρώ ότι θα πρέπει να εισαγάγουμε μέτρα που να έχουν κάποιο νόημα και αποτέλεσμα. Και, και στο τέλος επιτρέψτε να σημειώσω ότι η πρόταση αυτή για τη διάβρωση βάσης και μετατόπιση κερδών του ΩΣΑ πρέπει να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν για να έχουμε σωστά αποτελέσματα και να και να ικανοποιούμε το αίτημα και της κοινή γνώμη. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντοτε να αντιδρά μόνο όταν η κοινή γνώμη ασκεί πιέσει. Πρέπει πια να αρχίσουμε να διεκδικούμε την πρόοδο στην κατεύθυνση αυτή, να είμαστε πολύ πιο μπροστά από τις ε, πιέσεις της κοινή γνώμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Γουαλτιέρη, ο κύριος Χίλη, Συμφωνώ με το τελευταίο που είπατε ότι θα πρέπει να αντιδρούμε πριν τα παράπονα. Δεν θα επαναλάβω κάποια από τα επιχειρήματα που έχω ήδη εκφράσει, αλλά συμφωνώ με αυτό που είπατε για το κατεπήγον του θέματος, ότι πρέπει τέλος να ανασκουμποθούμε και να δράσουμε. Γιατί τώρα οι φορολογικές δικαιοδοσίες που δεν έχουν καλή διακυβέρνηση, ε, η φορολογική παράδειση δηλαδή. Γιατί μαύρη λίστα για αυτούς και γιατί όχι για όλους. Μπορούμε να έχουμε μια προσέγγιση όπου δημοσία... περιμένεις οι πολυεθνικές να δημοσιεύουν πληροφορίες για, φορολογικές, ε, για αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους ε, μόνο και όχι για τις υπόλοιπες φορολογικές δικαιοδοσίες. Η απάντηση είναι ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τη μελέτη αντικτύπου προκύπτει ότι ο ανταγωνιστικός κίνδυνος αποκάλυψης κάποιων πληροφοριών σε όλες τις τρίτες χώρες, δηλαδή ένας ανταγωνιστής μπορεί να δει σε αυτήν την περίπτωση ότι μια ευρωπαϊκή επιχείρηση συγκεντρώνει χρήματα το ώστε να κάνει επενδύσεις στην έρευνα και τεχνολογία ας πούμε, και προσλαμβάνει προσωπικό ούτως ώστε να επεκταθεί και σκέφτεται ας πούμε, να αγοράσει μια επιχείρηση, ας πούμε, να εξαγοράσει μια άλλη επιχείρηση. Όλε οι φορολογικέ δικαιοδοσίε θα έχουν περισσότερε πληροφορίε και μερικέ ε, εταιρείε μπορεί να φορολογηθούν διπλά σε αυτήν την περίπτωση. Σε περίπτωση μαύρη λίστα όμω, για του φορολογικού παραδείσου. είναι πολύ πιο δύσκολο νομίζω να επιχειρηματολογήσεις γιατί μια πολυεθνική συγκεντρώνει λεφτά σε ένα φορολογικό παράδεισο για επιχειρηματικούς σκοπούς. Μπορεί να είναι μόνο για φορολογικούς λόγους εκεί παρούσα και όχι για επιχειρηματικούς δηλαδή σκοπούς. Επίσης οι πληροφορίες που μπορεί να αποκαλυφθούν από τις δημοσίες πληροφοριών σε μαύρη λίστα μπορεί δεν μπορεί να δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια άλλη επιχείρηση. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει, ως μεσή γιατί συγκεντρώνεις λεφτά. Για επενδυτικούς σκοπούς ή για άλλους σκοπούς. Ο ανταγωνιστής σου δηλαδή μπορεί να καταλάβει. Επομένως πρέπει να κάνω αυτή τη διάκριση ανάμεσα στις τρίτες χώρες. Έχουμε γενικά τις τρίτες χώρες και έχουμε και μία μαύρη λίστα με φορολογικούς παραδείσους, γιατί αυτό που έδειξαν οι αποκαλύψεις του Παναμά είναι ότι μπορεί να κάνεις ερωτήσεις για κάποια θέματα, γιατί συμβαίνει σε αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους. Αυτό που ο κ. Μέσσερ Σμιτ για τη σχέση ανάμεσα σε αυτή την πρόταση για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στα έγγραφα του Παναμά που αφορούν περισσότερο εγκληματίες ας πούμε και διεφθαρμένους επιχειρηματίες αλλά και κάποιους έτσι που δρούν νόμιμα όμως σίγουρα. Γιατί αυτή η διάκριση λοιπόν, η απάντηση σε αυτό είναι ότι η δουλειά που κάνουμε στις εκθέσεις αναχώρα είναι πιο παλιά, πολύ πιο παλιά από τις αποκαλύψεις από τα έγγραφα του Παναμά. Είναι κάτι που μας έχει αποσχολήσει εδώ και καιρό, ας πούμε, και το θέλατε πολλοί από εσά να το κάνουμε. Δηλαδή εδώ και καιρό ασχολούμαστε με τις εκθέσεις αναχώρα. Η διαφορά με, τα, με τις αποκαλύψεις του Παναμά είναι ότι υπάρχει μια εστίαση τώρα στο θέμα αυτών των δικαιοδοσιών που δεν ε, σέβονται τους κανόνες για την καλή φορολογική governance και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να φτιάξουμε ένα, μια μαύρη λίστα και να επεκτείνουμε τις υποχρεώσεις υποβολή εκθέσεων, ειδικά για τις χώρες που είναι, για τις δικαιοδοσίε που είναι στο, στη μαύρη λίστα. Ε, εμείς ασχοληθήκαμε λοιπόν με τις εκθέσεις αναχώρα πολύ πριν το Παναμά. Απλώς τα έγγραφα του Παναμά μας δίνουν και μια άλλη διάσταση, Υπάρχει μια πλειά θέματων που αποκάλυψαν τα έγγραφα του Παναμά και με τα οποία ασχολείται ο κ. Μοσκοβισή. Η λίστα θα είναι έτοιμη εν ευθέτω χρόνο. Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία, ανυπομονησία στο γραφείο του Πιέα Μοσκοβισή. Θέλει να προχωρήσουμε Νομίζω ότι είναι πιο λογικό να προχωρήσουμε όπω θέλουμε εμεί, να κοιτάξουμε όλε τι δικαιοδοσίε, να εφαρμόσουμε τα κριτήρια, να δούμε ποιο τα σέβεται, ποιο δεν τα σέβεται, παρά να βάλουμε του πάντε ε, στη μαύρη λίστα και να έχουμε μια πολύ συγκρουσιακή κατάσταση. Ο στόχο νομίζω είναι πάντως αυτό Να εντοπίσουμε αυτού εναντίον των οποίων πρέπει να λάβουμε δράση. Τώρα, για τις κυρώσεις και την ε, εφαρμογή των κανόνων. οι κυρώσεις αναφέρονται στην οδηγία για τα λογιστικά. Την ευθύνη την έχουν τα κράτη-μέλη. Αυτά πρέπει να εφαρμόσουν την οδηγία. Πρέπει να είναι ε, αποτελεσματική, αναλογική, αποτρεπτική. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα επιβάλλουν τις κυρώσεις και θα καθορίσουν ποιες είναι αυτές οι κυρώσεις. Και μην ξεχνάτε τις ευρύτερες αποκαλύψεις που ακριβώς ε, είναι ένα επιχείρημα υπέρ της διαφάνειας. Πρέπει να υπάρχει δημόσιος έλεγχος. Ε, πρέπει να δούμε από την άλλη την επίπτωση στις επιχειρήσεις, ε, στους μετόχους, ε, στους καταναλωτές. και μπορεί να είναι πολύ σημαντικότερε από τι απλέ κυρώσει. Γιατί αν οι επενδυτέ, οι καταναλωτέ, ε, οι μέτοχοι φύγουν από μια εταιρεία, τότε αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να έχει τεράστιες επιπτώσεις. Μπορεί να είναι εντελώς ε, και απόλυτα ανατρεπτικό, πούμε, και συγκλονιστικό. Thank Σας ευχαριστώ. Περνούμε λοιπόν στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Πρώτος ο κύριος Καβαντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα τα πω πολύ γρήγορα. Χωρίς μικρόφωνο. Ένα τεχνικό ζήτημα προς τον Επίτροπο απευθύνομαι και ένα πολιτικό ουσιαστικά. που την ένθα πρέπει να διαχειριστούμε την οικονομία και τη φορολογία. Το τεχνικό ερώτημα είναι φορολογική βάση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό έδαφος πώς ε, θα υπολογιστεί με βάση το τζίρο, το κύκλο εργασιών, το καθαρό κέρδος πριν ε, την ενοποίηση ε, των κερδών σε μια εταιρεία holding. Αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό γιατί αυτό που αντικατοπτρίζει καλύτερα την οικονομική δραστηριότητα που κανονικά θα έπρεπε να υπόκειται σε φορολογία είναι ο κύκλος εργασιών, ο τζίρος. Δεύτερο, Κύριε Επίτροπε, δεύτερο ερώτημα απλό. Αν κατάλαβα καλά, δηλώσατε ότι η αρχή της οδηγίας αυτής θα είναι μια πολύ απλή έννοια. Δηλαδή, Οποιαδήποτε δραστηριότητα σε κάποια δικαιοδοσία, κάποια επιτράπη θα πρέπει να υποβάλλεται σε φορολογία ανεξαρτήτω ε, το αν πρόκειται για ευρωπαϊκή εταιρεία, για θηγατρική ευρωπαϊκή ή μη ευρωπαϊκή που κερδίζει χρήματα σε αυτή την επικράτεια. Δηλαδή υπάρχει η αρχή της φορολογικής αδαφικότητας, κερδίζω χρήματα σε ένα έδαφος, πληρώνω φόρους σε αυτό. Ευχαριστώ. Ράντεφ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση, την οποία στηρίζω, διότι ε, στηρίζω την ιδέα της μεγαλύτερης διαφάνειας για τη φορολόγηση των εταιριών. Ελπίζω δε ότι με τον τρόπο αυτό θα καλύψουμε κάποια κενά και κάποιες ασυμβατότητες μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων των κρατών μελών. Δεν έπρεπε να περιμένουμε το σκάνδαλο με τα έγγραφα του Παναμά για να κινητοποιηθούμε. Τώρα, το 2013, ο πρόεδρος ε, της ε, τότε Επιτροπής είχε πει ότι η χάνει ευρώ λόγω της ε, διαφθοράς και της, της απάτης μάλλον και της φοροδιαφυγής και βέβαια πλήττονται πιο πολύ από, αυτό, από αυτά διαφυγόντα κέρδη εθνική προϋπολογισμή. Με αυτές τις εκθέσεις αναχώρα την ερώτησή μου. μπορώ να καλύψω μια εταιρεία που κάποια παραρτήματά τη ή κάποιε θηγατρικέ δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκή επικράτεια και δεν συμμορφούνται οι δραστηριότητέ τη με τι απαιτήσει. Ποιος, ε, σε ποιον επιβάλλεται κυρώσεις, τι είδους κυρώσεις και ποιος ε, είναι ο αρμόδιος για τον έλεγχο, ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας. Επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η πρόταση, αλλά μένει πολύ δρόμος να εστιάσω σε κάποια ζητήματα. Το πρώτο φυσικά είναι το κατόφλι, συζητήθηκε διαμακρών. Δεν καταλαβαίνω όμως αν στόχος, όπως είπατε, είναι να έχουμε ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων και εθνικών αυστηρά επιχειρήσεων, δεν θα έπρεπε να προσπαθεί να καλύψει τον των περισσότερε πολυεθνικέ. Άρα θα ήταν πολύ πιο δικαιολογημένο ένα πιο χαμηλό κατόφλι για να ε, να καλύψετε έτσι τι περισσότερε πολυεθνικέ. Ε, Επίση, δεύτερο με πληροφόρηση. Εμεί έχουμε ζητήσει πάντοτε να έχουμε συγκεκριμένε πληροφορίε για επιδοτήσει, για ενεργετικό, για τι ε, ε θηγατρικέ. Είπαμε ότι όλα αυτά στοιχεία πρέπει να δημοσιοποιούνται από τι ε, εταιρείε για τι πολυεθνικέ. Γιατί περιορίζεστε σε τόσο λίγε πληροφορίε. Τρίτον, το οποίο το παν και άλλοι, συγκεκριμένες πληροφορίες κτλ. Δεν κατάλαβα πολύ καλά. Μας λέτε ότι δεν μπορείτε να επιβάλλετε τη δημοσιοποίηση σε όλες τις χώρες εκτός Ένωσης για τις πολυεθνικές που δεν είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Αλλά πώς τους επιβάλλετε σε κάποιες χώρες τουλάχιστον αυτή την υποχρέωση. Αφού μπορείτε να το κάνετε για κάποιες χώρες, μπορείτε να το κάνετε και για όλες τις άλλες. Εμείς αυτό θα προτιμούσαμε, φαντάζομαι, στη μεγάλη πλειοψηφία μας τουλάχιστον, δηλαδή να υπάρχει μέγιστη δυνατή διαφάνεια για όλα αυτά τα ερωτήματα και θέματα θα περιμέναμε πιο πολλά από την Κομισιόν. Πιο πολλά σημαίνει να ακολουθήσετε τη δική μας πρόταση που είχαμε προτείνει ως Κοινοβούλιο πολύ πιο φιλόδοξα πράγματα στην οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων και είχαν το τεράστιο πλεονέκτημα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πιο νωρίς και άλλα και στο χρονοδιάγραμμα θα ήμασταν πιο φιλόδοξοι. Σίγουρα ε, καλό θα ήταν ε, να μην ξεκινήσει εκ νέου μια νομοθετική διαδικασία ε, που θα είναι και πιο αδύναμη η αφιτηρία της και να συνεχίσουμε σε αυτή τη βάση αλλά βελτιώντας τα πράγματα. Ευχαριστώ και η τελευταία ερώτηση παρακαλώ από τον κύριο Μαρίνιο Πίντο. Επίτροπε. Οι αποκαλύψεις των γράφων του Παναμά εξέθεσαν τις διαστάσεις της παρανομίας που επιτρέπει να ξεφύγει κανείς από τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Και η ερώτηση που διατυπώνω προέρχεται από τον λαό που εκπροσωπώ. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση για να διορθώσει το πρόβλημα, πώς είναι δυνατόν να επιτρέπεται να υπάρχουν ακόμα υπεράκτιες πλατφόρμες offshore γιατί δεν υπάρχει πολιτική για να αντιμετωπιστούν αυτά τα παράνομα στα τελευταία ανάλυση συστήματα. Υπάρχουν επιχειρήσεις αποκλειστικά μάλιστα μέτρα στην Πορτογαλία που βλέπουμε όμως ε, να έχουν ε, τη φορολογική τους βάση στο Λουξεμβούργο ή και σε άλλες ε, χώρες. Γιατί λοιπόν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την, αυτό το αναθέμητο ανταγωνισμό τελικά μεταξύ των κρατών και γιατί δεν μπορούμε να επιβάλλουμε την αλληλεγγύη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ κρατών. Ευχαριστώ. Απάντηση. Καταρχάς, μια γενική παρατήρηση, μια και ερωτήθηκε αρκετές φορές. Γιατί χρειάστηκε να βγουν στη φόρα τα έγγραφα του Παναμά για να λάβουμε δράση, να ξεσπάσει το σκάνδαλο. Όχι, το ξαναείπα. Δεν περιμέναμε να δημοσιευθούν τα έγγραφα του Παναμά. Η πρόταση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο μέτρων όπου έχουμε την ε, ε, πρωτοκαθεδρία με τον κύριο Μοσκοβιστή και την κυρία Φεστάγκερ έχουμε, κάνει, έχουμε αναλάβει μέτρα πολύ νωρίτερα, έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό και νομίζω επίσης, και θα το επαναλάβω, ότι και τι αντιλαμβάνομαι βεβαίω τα επιχειρήματα ότι πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι και ότι πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω κτλ. Πιστεύω ότι είμαστε πιο φιλόδοξοι σε έναν βαθμό από ό,τι προηγούμενες προτάσεις, διότι ξεπερνούμε τις ε, καθαρά ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με την πρόταση αυτή και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία και για λόγους ανταγωνισμού. Έχει επίσης μεγάλη σημασία και για να αποσταλεί το μήνυμα ότι θέλουμε αυτές οι αρχές να ισχύουν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα μας λέτε ότι κάποιες από τις επιχειρήσεις που ενδεχομένως είναι οι πιο ε, πιθανές όπως θεωρούν οι ψηφοφόροι και ίσως και οι βουλευτές εδώ ε, οι πιο πιθανές να πληρώνουν λιγότερους φόρους νομίζω ότι εάν κάναμε μια πρόταση η οποία δεν κάλυπτε μη ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, δεν θα μπορούσε κανείς να καταλάβει αυτές τις επιλογές. Αυτό οδηγεί βέβαια σε άλλους παράγοντες, για τον τρόπο με τον οποίο εντετυπώσαμε την πρόταση, μπορεί να προξενούν δυσφορία αυτά που βλέπετε, αλλά καλύπτουμε, και αυτός είναι ο στόχος μας, καλύπτουμε όλες τις μεγάλες πολυεθνικές και όχι μόνο τις ευρωπαϊκές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συγκεκριμένε ερωτήσει τώρα που διατυπώθηκαν και μπορούμε τι λεπτομέρειε να τι συζητήσουμε και σε λίγο αν θέλετε τα τεχνικά ζητήματα δηλαδή τη φορολογική ε, βάση κτλ. Γιατί εδώ δεν προσδιορίζεται τη φορολογική βάση. Η βάση είναι αυτή που ορίζει το κράτος μέλος. Ο φόρος τον οποίο παραπέμπουμε είναι ο φόρος για επιχειρήσεις όπως ισχύει σε κάθε περίπτωση. Αλλά πολύ ευχαριστώ να συζητήσουμε σε λεπτομέρειες κάποια ζητήματα αν θέλετε να έρθετε να ζητήσω από το προσωπικό μου να έρθει σε επαφή μαζί σας. Γιατί λοιπόν δεν καλύπτουν πιο πολλές χώρες, το συζητήσαμε, γιατί δεν καλύπτουν πιο πολλές πληροφορίες. Έχουμε προσδιορίσει ε, μια κατηγορία πληροφοριών, ένα σύνολο πληροφοριών που θα είναι κοινέ θα διαβιβάζονται μεταξύ φορολογικών αρχών με βάση τις προτάσεις του ΟΣΑ. Και χάρη και στου δημοσιογράφου που κάνουν σχετικέ έρευνε, θα μπορούν οι πολίτες να ενημερώνονται, να διατυπώνουν τα ερωτήματα αν πράγματι αυτές οι επιχειρήσεις καταβάλουν φόρο στι χώρες στις οποίες αποκομίζουν, παράγουν το κέρδο του. Και νομίζω ότι ένα πληρέστερο κατάλογος πληροφοριών μάλλον αντίστροφα ένας κατάλογος με πιο ε, ασαφείς πληροφορίες μπορεί να αφήνει πολύ πιο διαυγή την εικόνα για ορισμένους από ότι ένας με πιο εξαντλητικές. Και νομίζω ότι είναι σωστή η επιλογή αυτή. Για δε τις κυρώσεις αυτές επαφήνται στα οικία κράτη-μέλη. Δεν προσδιορίζονται ποσά, όπως είπαμε, θα πρέπει να είναι αποτρεπτικές, αποτελεσματικές, αναλογικές οι κυρώσεις. Αλλά και όπως είπα και μόλις τώρα, το πιο αποτρεπτικό μέτρο είναι η αποκάλυψη στην κοινή γνώμη. Μια επιχείρηση η οποία δεν είναι σε θέση να εξηγήσει τι κάνει στο κοινό, στην κοινή γνώμη, προφανώς οδηγεί σε πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα και αυτό αποτελεί ένα ισχυρότατο μέτρο κύρωσης. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν ο χρόνος που είχαμε για την Επιτροπή των Οικονομικών. Ο κύριος Γκίγκολτ έχει το λόγο. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Σλιμ Μπέσερουγκ. Πολύ ωραία γερμανική λέξη. Ξέρετε τι θα πει. Όχι. Έτσι μια κακή μετάφραση είναι ε, βελτιώνω κάτι κάνοντα το χειρότερο. Αυτό θα πει αυτή η γερμανική λέξη. Και νομίζω ότι αυτό περιγράφει πολύ εύγλωτα την πρόταση που μας κάνατε, ε, αντιδρώντας και μάλιστα στα έγγραφα του Παναμά, αποκαλύψει αποκαλύψεις αυτές, διότι τώρα τελικά κάποιοι φορολογικοί παράδεισοι που έχουν μπει σε μαύρη λίστα, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν εκθέσεις και στα κράτη-μέλη της Ένωσης, για να αποφύγουμε υποτιθέμενα πλεονεκτήματα, μάλλον μειονεκτήματα, εάν επιβάλλουμε παντού στον κόσμο τέτοια πρότυπα για εκθέσεις αναχώρα. Αν θέλουμε να αποφύγουμε ε, κάποιες εταιρείες εκτός ένωσης ε, που δεν θέλουν να δηλώσουν, τελικά ε, νομίζω ότι εσείς με τις προτάσεις σας βλάπτετε την Ευρώπη ως ε, τόπο επενδύσεων. Γιατί θα ξέρουν εταιρείε που δραστηριοποιούνται τώρα σε διάφορε περιοχέ του πλανήτη ότι αν επενδύσουν στην Ευρώπη θα πρέπει να υποβάλουν εκθέσει, αν επενδύουν εκτό όχι. Άρα είναι κακή λύση αυτή που προτείνεται. Η μόνη πιστική λύση θα ήταν από ένα μέγεθος εταιρεία και μετά θα πρέπει να αναφέρονται τα κέρδη της εταιρεία ε, αναχώρα. Και αυτό να ισχύει οπουδήποτε στον κόσμο. Αυτή η διαφάνεια και μάλιστα ισότιμη διαφάνεια είναι η μόνη λύση γιατί καμία εταιρεία δεν θα έρθει στην Ευρώπη να επενδύσει αν πρέπει μετά να υποβάλει τέτοιε εκθέσεις. Αυτό είναι λοιπόν το Ferslim Besserung που, είπατε, αυτό που είπα. Αυτή είναι η, ε, ε, το να κάνουμε κάτι τελικά χειρότερο να θέλουμε να το βελτιώσουμε. ο μαύρος κατάλληλος αυτός τώρα ε, δεν θα λειτουργήσει και για έναν ακόμη λόγο, διότι οι πολιτικές πίεσεις στο παρελθόν δεν λειτουργήσαν και το ξέρουμε από τη ΣΥΠΑ που μπορεί κανείς να ανοίξει εταιρείε γραμματοκιβωτίου πάρα πολύ απλά ε, χωρίς να υπάρχουν αυτές οι κανόνες εκτισίας και από πολιτικές πλευρά είναι βάλτες αυτές οι μαύρε λίστε και πόσο τελικά ήταν αποτελεσματικέ οι κυβερνήσει. Κάποιο που είναι επιφυλακτικό στην πολιτική, μήπω πρέπει να πάει στην ε, αρχή τη ελεύθερη αγορά που λέει διαφάνεια για όλου και όχι να εμπιστεύεται την πολιτική για ένα παγκόσμιο μαύρο κατάλογο. Όπου είπα ποτέ δεν θα τολμήσει κανεί να. Τη δεν θα τολμήσει κανεί να τι βάλει εκεί είναι η πρότασή σα να βγει προς σωστή κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να γυρίσετε πίσω στην αρχική ιδέα και να σταματήσετε αυτέ τι ε, προσπάθειε Φερσλίν μπέσερου. και ελπίζω να έχετε μάθει πια αυτή τη λέξη μετά από τόσε φορέ που την είπα. Είμαστε και συνομοθέτε, βέβαια, έτσι, ε, λέει ο κ. Γκουαλτιέρη, άρα ε, να πω και σε εμά. Τώρα εμεί έχουμε στα χέρια μας αυτή την πρόταση, λέει ο κ. Γκουαλτιέρη. Μάρκο Τζάνι τώρα. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Και εγώ θεωρώ ότι η πρόταση αυτή δεν είναι πολύ φιλόδοξη, δεν είναι θαραλέα, γιατί σε μια τέτοια χρονική στιγμή μεγάλης πίεσης ε, πάνω στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να νομοθετήσουν προκειμένου να καταπολεμήσουν την φορολογική τη και φοροαποφυγή, νομίζω ότι υπολοιπόμεθα σε σχέση με τα όσα συμφώνησε ο Το Κοινοβούλιο έχει κάνει καλή δουλειά για κάποια νομοθετήματα. Πραγματικά θα πρέπει να βελτιωθεί η πρότασή σας, το πιστεύω αυτό. Σε ό,τι αφορά τα σημεία τα οποία είναι λιγάκι εκκρεμή, θα ήθελα να κάνω τις εξής ερωτήσεις. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το αίτημα και την υποχρέωση αποκάλυψης, μας εξηγήσατε πώς θα γίνει Δηλαδή θα γίνει βαθμιδόν καταρχάς και δεν θα βαραίνει πολύ τις επιχειρήσεις. Το να μην ζητάτε πληροφορίες, όπως παραδείγματο χάρη, ένα κατάλογο, ας πούμε, για το πού βρίσκονται οι θυγατρικές, να μην ξέρουμε από ποιες χώρες έχουν ληφθεί ε, δημόσιες ενισχύσεις, ε, πότε έχουν μετακινηθεί περιουσιακά στοιχεία ε, σε άλλες χώρες, ε, πότε έχουν γίνει πωλήσει κτλ. Αυτέ οι πληροφορίε είναι εκ των όνων κάνευ, ούτω ώστε αυτέ οι εκθέσει αναχώρα να είναι αποτελεσματικέ και να δίνουν τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Συμφωνώ με τι αμφιβολίε που εξέφρασε ο κύριο Γκίγκολτ μόλι τώρα. Δηλαδή, μία πρόταση που βασίζεται σε αυτέ τι προποθέσει, country by country reporting, μπορεί τελικά όντω να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό και να τιμωρήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μοναδική λύση για να εξασφαλίσουμε ότι οι εκθέσεις αυτές θα λειτουργούν και ότι δεν θα τιμωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το να έχουμε αυτή την προϋπόθεση για όλους και για όλες τις χώρες. Τελευταίο ερώτημα για αυτή τη βαθμιαία προσέγγιση που είπατε. Πιστεύετε ότι μία προνοιακή προσέγγιση... Συγγνώμη, συγγνώμη, ξεπεράσατε τα δύο λεφτά σας, λέει ο Πρόεδρος δεν θα δημιουργούσε μια καλύτερη, έτσι, ένα καλύτερο momentum. Η ε, κυρία Κάπελ και ευχαριστώ Επίτροπε. Έχει πάρα πολύ δουλειά για να καταπολεμήσει την φορά αποφυγή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει βέβαια να οδηγήσει περισσότερο προς μια αποτελεσματική φορολογία, να γίνεται δηλαδή φορολόγηση εκεί όπου υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα και βέβαια ισότιμε συνθήκε ανταγωνισμού. Δεύτερον, είπατε και εσεί ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει πληρώνουν πολύ βαρύτερο τίμημα φορολογικά από ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Και τρίτον, χρειάζεται διαφάνεια. Εδώ το country by country reporting είναι ένα πολύ καλό βήμα για τη διαφάνεια. Οι πολυεθνικές συγκεκριμένες επιχειρήσεις με 750 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα πρέπει να δημοσιοποιούν τους, τα κέρδη τους και τους φόρους εκεί που τους πληρώνουν. Αυτό θα, και θα πρέπει να τους καταβάλουν σε κάθε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, τα πράγματα αλλάζουν λίγο μετά την δημοσίευση των αγραφών του Παναμά, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν φορολογικές ε, περιφέρειες, περιοχές όπου δεν ισχύει η φορολογική νομοθεσία, η φορολογική παράδειση θα λέγαμε και χάρη σε αυτούς μπορούν να αποφύγουν τη φορολογία οι εταιρείε. Βεβαίω. οι βέλτιστες πρακτικές που προσπαθούν, που τίνουν προς την ε, δέσμευση περισσότερο και με το country by country reporting και που έχουμε και από οργανισμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα, ο και ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών ε, προωθούνται και νομίζω ότι έτσι μπορώ να φτάσω στην ερώτησή μου. Σε ένα έγγραφο εργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται λόγο για πιο αυστηρή στάση απέναντι σε τράπεζε και φοροτεχνικού. Γιατί λέει τα έγγραφα του Παναμά δείχνουν ότι οι φοροτεχνικοί και οι τράπεζες έχουν ενεργώ υποστηρίξει τους πελάτες του ω προς την διαδικασία που οδηγεί στην φόρο αποφυγή, θα υπάρξουν μέτρα, λέει, αποτροπής. Τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα, είναι η ερώτησή μου. Ποια είναι αυτά τα μέτρα αποτροπής και μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες. Ευχαριστώ και μπορούμε να δώσουμε από ένα λεπτό σε δύο κατστιά. Η Σάλβα και Τάνι. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Συμφωνούμε λοιπόν όλοι. Φαντάζομαι ότι έχουν πια μπουχτίσει οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο και νομίζω ότι θα πρέπει να δουλέψετε κύριε Επίτροπε για την υλοποίηση των προτάσεων το ταχύτερο δυνατό. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι τράπεζες πρέπει να κάνουν τις εκθέσεις αναχώρα και αν δεν το πράξουν αυτό δεν θα καταλάβει ο πολίτης γιατί αυτές οι επιχειρήσεις δεν προβαίνουν σε εκθέσεις αναχώρα. Και αυτό είναι και το επιχείρημά μου και ένας λόγος παραπάνω πρέπει να υποχρεωθούν, να καταστεί υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις να ε, πραγματοποιούν και να δημοσιεύουν τις εκθέσεις χώρα. και θέλω τη γνώμη σας κύριε Επίτροπε. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κύριο Στάνγκ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ξεκινώ λέγοντας ότι έχει κρίσιμη σημασία αυτό το νομοθέτημα με τα έγγραφα του Παναμά είδαμε ότι η διαφάνεια έχει κέρια σημασία για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Κάθε πρωτοβουλία λοιπόν που λαμβάναν λαμβάνεται προς την κατεύθυνση αυτή θα είναι ένα ακόμα βήμα και το μοναδικ... η μοναδική λύση για να κερδίσουμε γιατί πάντα θα είναι συνεχής ο αγώνας βέβαια θα προσπαθούν οι φοροδιαφεύγοντες να αποφεύγουν την καταβολή των φόρων αλλά με την δημοσιοποίηση μπορούμε να κερδίσουμε πολλά. Δύο ερωτήσεις λοιπόν γιατί δεν είναι σαφές για μένα Μιλάτε για μια μαύρη λίστα εσείς και υπάρχει και μια μαύρη λίστα στο, στο πακέτο για την αποφυγή, για τη φοροαποφυγή, για την καταπολέμηση φοροαποφυγής. Ε, ο, η ίδια μαύρη λίστα είναι νέου ναι και πώς μπορούν ε, να υποχρεωθούν ε, και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε country by country reporting. Δεύτερον, μπορεί να υπάρχει πάνω από μια δικαιοδοσία, όπως ξέρετε, συμβαίνει στις κάτω και στη δική σας τη χώρα, μέσα στην ίδια κρατική επικράτεια διαφορετικές δικαιοδοσίες. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να ζητήσουμε αναλυτικά και όχι ενοποιημένα στοιχεία και αναλόγως της φορολογικής δικαιοδοσίας μέσα στην ίδια κρατική οντότητα. Ο Επίτροπος. Υπάρχει αυτό το ερώτημα που επανέρχεται γιατί να μην έχουμε τους ίδιους κανόνες παντού, πώς θα εξασφαλίσουμε την ισότιμη μεταχείριση. Συμφωνώ απολύτως ότι σε έναν ιδανικό κόσμο θα είχαμε ένα σύστημα που θα ίσχυε διεθνώ ισοτίμος δικαίως και στα πλαίσια της πρόοδου που σημειώνεται εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από τον ΩΣΑ και από άλλους, Έχουμε φτιάξει μια διεθνή συνένεση και όλοι πιστεύουμε στην αρχή της διαδικασίας ότι θα το πετυχαίναμε αυτό. Αυτό ακριβώς. Το πρακτικό όμως πρόβλημα στο οποίο προσκρούμε είναι ότι αν δεν μπορείς να υποχρεώσεις όλες τις τρίτες χώρες να προσεγγίσουν τα πράγματα με τον δικό μας τρόπο, κινδυνεύεις να βρεθείς ενώπιον κάποιον από, από τα προβλήματα που συζητάμε. Έχω ήδη δει στο παρελθόν, στο μέτρο ε, για την υποβολή εκθέσεων της εξορρυπτικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας ξυλίας, ε, Είχαμε πείσει στι ΗΠΑ να υποχρεώσουν ε, αυτές τις ε, βιομηχανίες να υποβάλουν στοιχεία. Ακόμα δεν το έχουν κάνει. Θέλαμε κάτι που να αφορά όλους. Και τώρα το θέλουμε, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε τα εμπόδια στα οποία προσκρούμε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε υποβάλει αυτό που υποβάλαμε, που κατά την άποψή μου είναι ισορροπημένο κείμενο, ισορροπημένη προσέγγιση. Πιστεύω ότι για τις υποχρεώσεις ε, δημοσίευσης και αποκάλυψης στοιχείων, η προσέγγιση μας είναι τολμηρή. Καταλαβαίνω απόλυτα βέβαια ότι κάποιοι από εσάς θα θέλατε κάτι παραπάνω. Αλλά με το να εφαρμόσουμε αυτά που εφαρμόζουμε και σε μη ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και στι θηγατρικέ του μέσω των θηγατρικών, με το να πάμε πιο πέρα από εκεί που έφτασε ο ΩΣΑ, με το να έχουμε όλε αυτέ τι υποχρεώσει για την υποβολή εκθέσεων. Είμαστε η πρώτη δικαιοδοσία ή θα είμαστε, ελπίζω, το συντομότερο δυνατόν, να πετύχουμε αυτά τα πράγματα. Επομένω είμαστε τολμηροί. Αλλά ακούω πολλοί από εσά να λέτε ότι θέλατε κάτι παραπάνω. Τώρα για το συγκεκριμένο ερώτημα το μέτρο που μπορούμε να λάβουμε για τις τράπεζες και τους ε, χρηματοπιστωτικούς συμβούλους. Οι χρηματοπιστωτικοί σύμβουλοι που μπορεί να δίνουν συμβουλές σε εταιρείε για να προωθήσουν κλιματικές δραστηριότητε. Φυσικά αυτό είναι ένα τομέας που ερευνούμε. Έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια, αλλά δεν μπορώ να σας πω σήμερα τι μέτρα θα πάρουμε. Αλλά ασχολείται με το θέμα αυτό η Κομισιόν. Έχουμε τέτοιο καθεστώς για την κατάχρηση της θέσης στην αγορά με εγκληματικό τρόπο, αλλά θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να εφαρμόσουμε κάτι τέτοιο και σε άλλους τομείς. Συμφωνώ αυτό που είπατε, ότι με τις υποχρεώσεις περί εκθέσεων για τις τράπεζες πετύχαμε μεγαλύτερη διαφάνεια και αυτό είναι ένα ε, πολύ σημαντικό εργαλείο. Συμφωνώ απόλυτα ότι αυτό χρειαζόμαστε γενικά να το εφαρμόσουμε όχι μόνο στις τράπεζες, ε, όχι μόνο στην εξωτερική βιομηχανία, αλλά σε όλες τις μεγάλες ε, πολυεθνικές. Όχι μόνο στις ευρωπαϊκές τράπεζες και στις άλλες, στις ξένες, ευρωπαϊκές, στις ξένες τράπεζες που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις ε, εκθέσεις ε, αναδικαιοδοσία. Είναι εκτός του χαρτοφυλακίου μου. Θα το διαβάσω το θέμα αυτό στον Πιέρ Μοσκοβισή που έχει μια εντολή ε, πολύ πιο ευρεία από τη δική μου. Υπάρχουν διάφορα θέματα που προέκυψαν από τις αποκαλύψεις του Παναμά για επιμέρους κράτη-μέλη. Είδαμε ότι διάφορα κράτη-μέλη κάνουν προτάσεις για τις προτεραιότητε δράσης. Είναι η απαρχή της συζήτηση αυτή εδώ. Που... Και θα συνεχίσει σίγουρα αυτή η συζήτηση και με τη συμμετοχή των Ευρωβουλευτών και του κοινού εν γέννη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. να ευχαριστήσω τους Προέδρους των τριών επιτροπών. Ε, σίγουρα θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερο χρόνο να αφιερώσουμε στη συζήτηση του πολύ σοβαρού θέματος, αλλά είναι όλων ο χρόνος περιορισμένος. Σας ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε στο άμεσο μέλλον να έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε μαζί σας.